mercosur μπορεί να υπονομευτεί στην πράξη. μπορεί στην πραγματικότητα η βραζιλία να αποχωρήσει από, το κλίμα, από τη συμφωνία του κλίματος για το πορίσι. μπορεί στην πραγματικότητα η βραζιλία να αποτελέσει την αιτία του ναυαγίου. Sorry, we really have to get... Συγγνώμη, πρέπει να προχωρήσουμε. Next... Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Γιον Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο Τραμπ ε, τον ΠΟΕ ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να θέλει άτακτο Brexit και η Ευρώπη πλήττεται. Ε, είμαστε η μεγαλύτερη αγορά από πλευράς καταναλωτών. Έχουμε μεγάλη ευθύνη αλλά και ευκαιρία ε, για να γίνει βιώσιμη η ε, ανάπτυξη και το εμπόριο θα πρέπει εμείς να ηγηθούμε. Η Πράσινη Συμφωνία ζητάει δράση μπορούμε και οφείλουμε στο μέλλον σε εμπορικέ συμφωνίε, να ορίζουμε ότι πρέπει να τηρείται η Συμφωνία των Παρισίων και να μπορούν και να επιβάλλονται και ε, οι αντίστοιχε κυρώσει. Και θα πρέπει να τα εφαρμόζουν και οι Κινέζοι και ο Μπολσονάρο και ο Τζόνσον και ο Τραμπ. Δεν μπορεί ένας κλιματοσκεπτικιστής να τα στυλώνει στη Μαδρίτη και να καταστρέφει τον Αμαζόνιο. Δεν είναι καλός εταίρος αυτός εμπορικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο θα είχε η κυρία Βάης κανονικά, την οποία όμως δεν βλέπω ε, στο ημικύκλιο. Η κυρία Βάης, δεν τη βλέπω. Ε, προχωρούμε. Η κυρία Πιετικάινεν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ε, ε, μελετούμε τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, τις παλαιότερες και τις καινούριες. Ε, όπως αυτή που μας απασχολεί αυτό τον καιρό, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τις χώρες Μερκοσούρ. Ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και καταπολεμά την κλιματική αλλαγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ε, απεμπολίσουμε τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με συμφωνίες παλαιού τύπου. Θα πρέπει τώρα να έχουμε σύγχρονες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών γιατί έχει τεράστιες επιπτώσεις αυτό για τους εργαζομένους, για τις διαδικασίες παραγωγής, ε, για τη δική μας παραγωγή τροφίμων κλπ. Ζωική πρόέλευση για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στα ζώα, για τον ε, ε, τρόπο με τον οποίο παράγουμε σόγια και τι σημαίνει αυτό για τα δάση στον Αμαζόνιο. Οι συμφωνίε αυτέ λοιπόν ελευθέρων συναλλαγών δεν μπορούν να επικεντρώνονται μόνο στα οικονομικά ζητήματα και στα εμπορικά. Η κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τη Μερκοσούρ έχει στο περιεχόμενο της κάποιους όρους ε, που ε, συνηγορούν στο να υιοθετηθούν συγκεκριμένα κοινωνικά στάνταρ. Επίσης μπορούμε να περάσουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Όμως έχει και ένα ρίσκο αυτή η συμφωνία. Έχει ε, μια αρνητική επιρροή στην γεωργία. Ο κύριος ε, Χόγκαν έχει υποσχεθεί κάποιο δισευρό στους γεωργούς μας ε, και όμως ε, αυτή η συμφωνία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή, όμως ο κύριος Μπολσονάρο δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι και να, ερημώνει, να περιμώνει την Αμαζονία. Νομίζω ότι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Μερκοσούρ είναι αποδεκτή μόνο εάν ο Μπολσονάρο εγγυηθεί με συγκεκριμένα μέτρα ότι θα σταματήσει την αποψήλωση και την παράνομη υλοτομία. Μόνο με αυτή την απτή εγγύηση του Προέδρου Μπολσονάρο ε, μπορούμε να ε, ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Επίσης πρέπει να δούμε πώς οι στόχοι οι συμφωνίες για το κλίμα μπορούν να αυξηθούν. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφο ε, Φερνάντε ε, για 1,5 λεπτό είναι ο τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συμφωνία με τι χώρε Μερκοσούρ είναι κάτι περισσότερο από την οικονομία. Είναι και αξίε, είναι βιώσιμη ανάπτυξη, είναι κοινωνική συμβασμή και βιωσιμότητα ε, στην απέτηση για αμεβιότητα καθώ και συμβατότητα με την ε, Πράσινη Συμφωνία για τα κολλικά τη Ευρώπη. Είναι μια τέλεια ευκαιρία που δεν μπορούμε να την ε, χάσουμε. Μέσα από τη συμφωνία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε Μερκοσούρ δεσμεύονται να υλοποιήσουν στην πράξη τη Συμφωνία των Παρισίων. Η συμφωνία με τι χώρε Μερκοσούρ ε, περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία των δασών, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών. Επίσης, δίνει φωνή στην κοινωνία των πολιτών, διότι υπάρχει και μηχανισμός για την παρακολούθηση της υλοποίησης της συμφωνίας και προβλέπει την προστασία των δικαιωμάτων των πληθυσμών ηθαγενών. Επίσης, περιλαμβάνει και την αρχή της προφύλαξης από τους πλέον καινοτόμους μηχανισμούς για να καταπολεμηθούν οι κλιματικές αλλαγές. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι η συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ είναι κάτι που θα φέρει σταθερότητα και στις εσωτερικές σχέσεις των ε, χωρών της Λατινικής Αμερικής όταν εγκριθεί. Δεν πρέπει λοιπόν να τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν πρέπει να πάει χαμένη αυτή η πρόταση. Είναι απολύτως συμβατή και θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα. Να συμβαδίσει με την Πράσινη Συμφωνία το New Green Deal. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην Επιτροπή, ο Επίτροπος κ. Χόγκαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους 64 ομιλητές που συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο νέος φακός μέσα από τον οποίο τόσες πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές ε, θα πρέπει ε, να εξετάζονται πλέον. Πραγματικά το Πράσινο ε, Κόμμα είπε πολλά πράγματα υπέρ της Επιτροπής Φοντερ Λάιεν και το τι πρέπει να κάνει για την Πράσινη Συμφωνία. Αλήθεια, γιατί δεν ψηφίσατε την κυρία Φαντερ Λάιεν στην ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία μάλλον. Ποτέ μάλλον δεν είστε ικανοποιημένοι. Να συμφωνήσω με τον κύριο Γιουγκέρους, ο οποίος είπε, κυρία Γιουγκέρους, ο οποίος είπε ότι είναι ε, συμφωνή η ευκαιρία μας σήμερα ε, δεν έχουμε καν συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ για να βρούμε έναν τρόπο αυτές οι τέσσερις χώρες ε, να αγκαλιάσουν μια πιο προοδευτική ευκαιρία για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Πολλές από τις ανησυχίες που ανέφεραν μέλη εδώ του Κοινοβουλίου Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω άλλο μηχανισμό πέραν της επιστολής ή του να μιλάμε στο κοινοβούλιο ή στα διεθνή φόρα. Δεν ξέρω άλλον μηχανισμό ε, κινητοποίηση πέραν των, ε, ρυθμίσεων, των εμπορικών ρυθμίσεων. Οπότε σίγουρα για μένα είναι μια ευκαιρία αυτέ οι χώρε να μπουν στο παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί ομιλητέ εδώ μέσα που δεν έχουν εξετάσει τη συμφωνία. Του λέω με σεβασμό λοιπόν να την ξανακοιτάξουν και να κάνω και κάποιε παρατηρήσει. Ε, το να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μερκοσούρ είναι υπεύθυνη για τις φωτιές στον Αμαζόνιο και να περνάμε τέτοια μηνύματα στις χώρες είναι βλακεία ο, όντως αυτό που κάνει ο πρόεδρος Μπολσονάρο είναι φρικιαστικό. Έχει ε, τελείως αγνοήσει τον Αμαζόνιο. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Όμως ε, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σενάριο δεν θα ξανασυμβεί. Τι περιθώρια έχουμε να τον κινητοποιήσουμε ώστε αυτός και η κυβέρνησή του να προστατέψουν αυτό το υπέροχο θαύμα της φύσης. Ε, όλοι μας ε, το, συμμεριζόμαστε αυτό το στόχο. Η συμφωνία είναι σίγουρα μία συμφωνία η οποία εδώ και 20 χρόνια έχει τύχει διαπραγμάτευσης. Τελικά έχουμε βρει μία βάση για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπημένη σχέση με στόχο τη βιωσιμότητα. Ο πρόεδρος ε, Μπολσονάρο έκανε εκστρατεία ε, προεκλογικά λέγοντας ότι δεν θέλει να είναι στη Συμφωνία των Παρισίων. Είχε ακριβώς την ίδια θέση με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά άλλαξε γνώμη μέσα στα πλαίσια αυτή τη συμφωνία. Και τώρα έχει αγκαλιάσει τη συμφωνία των Παρισιών. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει ως προς την εφαρμογή όμως να πω στους ανθρώπους που λένε ότι δεν έχει γίνει πρόοδος για τη βιωσιμότητα, ότι υπάρχει μια δεσμευτική ρήτρα ε, για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισίου. Όλες οι χώρες που υπογράφουν ε, πρέπει να την τηρήσουν. Η Βραζιλία έχει ε, υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα για το 2030. Μηδέν παράνομη αποψήλωση στον Αμαζόνιο και αποζημίωση για τις εκπομπές δεξιδίου του άνθρακα. Δεύτερον, αποκατάσταση των δασών, 20 εκατομμύρια εκτάρια ε, πρέπει να αποκατασταθούν. Πλήρης εφαρμογή του κώδικα για τα δάση, ε, διατήρηση των φυσικών δασών και πάυση των παράνομων μη βιώσιμων πρακτικών. 20 εκατομμύρια εκτάρια μέχρι το 2030 είναι ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο σε σχέση με το μισό εκατομμύριο που αποψηλώνεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, πώς θα έχουμε τις δεσμεύσεις που θέλουμε Πραγματικά αναρωτιέμαι, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Η συμφωνία αυτή θα είναι επίσης ένα ισχυρό πλαίσιο για να έχουμε διατάξεις σχετικά με τους ηθαγενείς πληθυσμούς και τις βιώσιμες αλυσίδε τροφοδοσίας. Η συνεργασία για πιο βιώσιμα κοινωνικά προϊόντα που θα εμπλέκουν αυτές τις κοινωνίες είναι σημαντική. Μην λέτε λοιπόν ότι τους αγνοούμε. Για τα κοινωνικά δικαιώματα που είπαν πολλοί ομιλητές, όλες οι χώρες της Μερκοσούρ έχουν ε, κυρώσει τις ε, συμβάσεις του ΆΕΛΟ. εκτός από μία, σε μία χώρα. Τρεις χώρες λοιπόν έχουν κυρώσει και μία δεν έχει ε, κυρώσει μία συμφωνία. Πώς λέτε λοιπόν ότι δεν έχουμε κάνει κοινωνική πρόοδο και αυτό είναι λάθος. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μερκοσούρ έχουν ε, διαπραγματευτεί και τις εργασιακές διατάξεις Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε κοινή υποστήριξη, να υπάρχει κοινωνική πρόοδος ε, και ανάπτυξη. Η συμφωνία αυτή λοιπόν θα έχει μια ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ε, και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συγκεκριμένες συμβάσεις, σωστές ώρες εργασίας. Αυτά είναι παραδείγματα που δεν αναφέρθηκαν στη συζήτηση αλλά είναι στη συμφωνία. Πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη συμφωνία ε, πιο καλά. Εντάξει, τα αγροτικά προϊόντα, όπως α πούμε η ζάχαρη, είναι πολύ ε, ευαίσθητα και γι' αυτό έχουμε δασμούς. Έχουμε Έχουμε 276.000 τόνους εμπόριο με τη Μερκοσούρ ήδη ε, και δεν έχουμε ε, όρους ε, που να πληρούνται γιατί τα ευρωπαϊκά στάνταρ δεν τηρούνται και δεν μπορούν οι χώρε του Μερκοσούρ να τα τηρήσουν. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να έρθει εδώ χωρίς αυτά τα στάνταρ, ειδικά γεωργικά, αν δεν γίνουν 100% έλεγχοι. Ο λόγος λοιπόν που πολλά προϊόντα επιστρέφονται στι χώρε είναι ότι λειτουργούν οι έλεγχοι. Έχουμε 100% ελέγχους τη στιγμή. Και αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μου να συνεχιστεί. Δεν θα υπάρξει μείωση των στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα προστατεύσουμε όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις. Θα προστατευτούν. Υπάρχει μια ε, σφραγίδα ποιότητας. Ε, ξέρετε ότι ειδικά στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία αυτά ε, τιμούνται ιδιαίτερα. κύριε Γουάλλας, να από ότι ενδιαφέρεστε πολύ για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και το χαιρετίζω. Όμω, να σας εξηγήσω καλέ μου φίλε, τι μεγάλες πρόοδοι έχουν γίνει στο περιβάλλον και στην κοινωνική προστασία. Ε, αυτό θα σας ε, καθησυχάσει και θα μπορείτε να πείτε στην εκλογική σας περιφέρεια πώς γίνονται όλα αυτά. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποιο μοχλό για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι περιβαλλοντικέ οικονομικέ και κοινωνικές διαστάσεις ε, των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου χρησιμοποιούνται. Όπως είπαμε στη συζήτηση, ε, χρειάζεται μία διαδικασία ε, εξέτασης που θα μας δείξει πώς θα βελτιώσουμε τη συμφωνία και, να, ε, και θα αντικατοπτρίσουμε τις ανησυχίες ε, των μελών. Η ερμηνεία της συμφωνίας και οι διασαφήσεις που ζητήσατε θα σας δοθούν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προοπτική έγκριση αυτής της συμφωνίας. Πρέπει να εγκρίνει και να δώσει τη συνένεση του το σώμα πριν πάμε στα κράτη-μέλη. 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε διαπραγματεύσεις με τους φίλους μας στη Λατινική Αμερική προσπαθούσε να χτίσει τα, ε, τους δεσμούς που τόσα χρόνια τους αγνοούσαμε. Ήρθε η στιγμή λοιπόν ε, να ε, δείξουμε σε αυτούς τους φίλους μας ότι θέλουμε να περπατήσουμε χέρι-χέρι μαζί τους σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ Επίτροπε κύριο Γουάλλας, ε, αν είχε την ε, δικαίωμα να δείξει μπλε κάρτα τώρα στον Επίτροπο, θα του άρεσε πολύ, αλλά πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο, στο κυρία του Πουκράινεν. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επίκαιρη και χρήσιμη συζήτηση. Και το θέμα αυτό ανησυχεί όλου μα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύτιμα σχόλιά σας. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είχατε να πείτε και θα τα διαβιβάσω σίγουρα στο Συμβούλιο. Όλοι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και άλλα τέτοια ζητήματα και προβλήματα που είναι όλο και πιο επίγοντα. Η νέα πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει μια συνολική στρατηγική την οποία θα χρειαστούμε όλοι για να τη μελετήσουμε σε βάθος. Καλώς ορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τον Επίτροπο Χόγκαν γι' αυτό. Το εμπόριο συνιστά ένα σημαντικό τομέα πολιτικής, ε, όπου η βιωσιμότητα είναι ουσιαστικό στοιχείο. Είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας με τους εταίρους μας για το κλίμα και την περιβαλλοντική δράση και η Συμφωνία Μερκοσούρ υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ειδωθεί ως ευκαιρία για να προωθήσουμε αλλαγές. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα, ως ευκαιρία για να προωθήσουμε αλλαγές. Και αυτό δεν θα γίνει από μόνο του. Ορισμένοι από εσά αναφερθήκατε στην δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης, καλύτερης συμφωνίας. Αγαπητοί φίλοι, τώρα είναι πιο εύκολο να το λες αυτό παρά να το κάνεις. Η τρέχουσα συμφωνία μπορεί να μην είναι τέλεια, που δεν είναι ποτέ καμία συμφωνία. Οικονομικά όμως έχει μεγάλη σημασία και είναι επίσης μεγάλη πολιτική και η γεωπολιτική συμφωνία που υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο Μερκοσούρ και κατά τα άλλα αποτελεί και μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξάγει ψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Δεν μπορεί από μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει και να αναχαιτήσει την αποψήλωση των δασών. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Και ισχύει και για τις εμπορικές συμφωνίες και ιδιαίτερα τα κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αγαπητοί φίλοι, πιστεύω λοιπόν ότι το εμπόριο μας προσφέρει ε, πραγματικά δυνατότητες μόχλευσης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε και να δεχθούμε ότι αυτό αναπόφευκτα τελικά θα έχει και κάποια ανταλλάγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνεται εδώ η παρούσα συζήτηση. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής για την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα. China εδώ μπορείτε να ζητήσετε το λόγο στο Catch the Eye με το παραδοσιακό τρόπο ή και με τον ηλεκτρονικό. Και για τη γαλάζια κάρτα ισχύει Περιμένουμε λίγο να καθίσουν οι επίτροποι και θέλω να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας και να τους πω ότι δεν υπάρχει τείχος ανάμεσά σας και ανάμεσά μας και επειδή έχετε ακουστικά και δεν ακούτε και θέλετε να μιλάτε με τους διπλανούς σας ε, δεν ακούτε ότι κάνετε θόρυβο και ακούγεται γιατί ε, ακούγεται πάρα πολύ κάτω. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μην μιλάτε. Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας. Θα δώσω το λόγο τώρα ε, στον κύριο Μπορέλη τον οποίο και καλωσορίζω. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένα έχει συζητήσει την κατάσταση στην Τζιν ε, και διμερός στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και ε, πρόσφατα το έθεσα υπόψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Ανησυχούμε βαθύτατα και εξακολουθούμε για την κατάσταση στα στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και αυτό αφορά περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Άλλη μεγάλη πηγή ανησυχία είναι η χρήση ε, της πολύ δυσδυτική παρακολούθησης. Νέες τεχνολογίες με βιομετρικά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη παρακολουθούν τον κόσμο στην περιοχή Xinjiang, ε, στην αυτόνομη αυτή περιφέρεια, με βιομετρικά δεδομένα και με ευρεία κλίμακας αναγνώριση προσώπου, χαρακτηριστικών του προσώπου. Και πραγματικά ε, εδώ είναι ένα θέμα εθνότητα και θρησκείας ε, από χώρο λατρείας και περιορισμό στην ε, θρησκευτική εκπαίδευση και σε γλώσσες μειονοτήτων. Βεβαίως κάθε χώρα ε, έχει δικαίωμα να προχωρεί σε θεμητά μέτρα για να καταπολεμά την τρομοκρατία. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά η καταστολή και η αστυνομοκρατία στο Τζιντζάνγκ είναι δυσανάλογη με την αντίστοιχη προσπάθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα Ηνωμένα Έθνη ε, ε, ανέλησαν την αντιτρομοκρατική πολιτική της Κίνας και ανησυχούν βαθύτατα για τις ε, διαδικασίες αυτές και την έλλειψη δικαστικής εποπτείας. Θα ήθελα επίσης ε, να έχουν ανεξάρτητοι παρατηρητές απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή όπως η ε, ειδική εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών και η ύπατη εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι τώρα αυτές οι εκκλήσεις είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ε, θα ήταν σημαντικό βήμα να το δεχτούν. Το έχω θέσει υπόψη των Κινέζων αυτών και των πρέσβων. Ε, θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε μια τέτοια επίσκεψη εκεί. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη θρησκεία και στην άσκηση της λατρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να διατρανώνει αυτή τη θέση αρχής και να εκφράζει τις ανησυχίες για το Xinjiang στον πολιτικό διάλογο με την Κίνα και διεθνώς και φυσικά και στα Ηνωμένα Έθνη. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσω να ε, απευθύνω έκκληση στην Κίνα να ανταποκρίνεται στι εθνικέ και διεθνεί υποχρεώσει τη και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Κυρία Πρόεδρε, ε, ε, αγαπητοί βουλευτές, περιμένω με χαρά τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Βίζελερ Λίμα έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, εδώ και 20 χρόνια η Κίνα έχει συνάψει το Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά δικαιώματα για τα δικαιώματα των πολιτών. Έκτοτε η Παγκόσμια Επιτροπή περιμένει να το κυρώσει. Η Κίνα έχει επιτελέσει πρόοδο στον τομέα των κοινωνικών θεμάτων, αλλά τα πολιτικά δικαιώματα διαρκώς υποβαθμίζονται. Συλλήψεις, φυλακίσεις, ε, κατάργηση δικαιωμάτων ολόκληρων κοινοτήτων, όπως ε, αυτά των Ουιγούρων στην περιοχή της ε, Ξινιάνγκ. Το κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει αδρανές μετά τις αποκαλύψεις των China Cables. Οι πιέσεις κατά των Ουιγούρων είναι τεράστιες και συστηματικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής και οι αντιδράσεις μας δεν θα πρέπει να μείνουν στα λόγια, αλλά θα πρέπει να αναλυφθούν ευθύνε από τους αρμοδίους. Βραβεύσαμε τον τότε με το βραβείο Ζαχάροφ και αυτό είναι μια σαφής έκφραση του πώς βραβεύεται η ειρηνική μάχη για τα δικαιώματα μιας ε, ολόκληρης ομάδας του πληθυσμού και πώς κάποιος φυλακίζεται βεβαίως απλώς γιατί ζητά το δικαίωμα να έχει φωνή ο λαός του. Ε, είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν ε, με τους Ιγούρους στην περιοχή της Ξενγιάνγκ για ένα μεγάλο έθνος του 21ου αιώνα. Οι άνθρωποι αυτοί στους ε, καταπλησμούς, στα στατόπεδα αυτά επανεκπαίδευσης, λένε οι Κινέζοι, είναι οικειοθελείς και τα χαρακτηρίζουν σχεδόν οικοτροφία. Εδώ ε, η Κίνα θα πρέπει να επιτρέψει σε δυνητής παρατηρητές και δημοσιογράφους να ε, θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν εθνικά και να ζήσουν τις θρησκευτικέ τους πεπιθήσεις ελεύθερα. Ε, είναι επίσης απαραίτητο στα μάτια μου να παρακολουθούμε το, τα προϊόντα που παράγονται στα ζωτόπεδα αυτά να μην διατίθενται στα, στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία εταιρεία, καμία επιχείρηση να μην δέχεται να υποφελείται από την ε, καταναγκαστική εργασία. Ο καθένας, τα καταναγκαστικά έργα. Θα πρέπει ο καθένας εδώ να αναλάβει τις ευθύνες του. Ευχαριστώ. Ε, εδώ η κυρία Πύρη τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μπορέλ. Πρώτα απ' όλα σα καλωσορίζουμε θερμά από το Ευρωκοινοβούλιο και εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στι νέε σα αρμοδιότητε σα συγχαίρουμε. Θέλουμε στενή συνεργασία για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα είναι ένα από του σημαντικότερου εταίρου τη Ένωσή μα και είναι ένα κεντρικό μέλο τη διεθνού κοινότητα. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εθελοτυφλούμε στι σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνω από ένα εκατομμύριο Ιγούροι και καζάκι. Ε, είναι φυλακισμένοι Χωρί να έχουν δικαστεί, χωρί κατηγορίε. πολύ απλά γιατί είναι μουσουλμάνοι, χωρί κανένα λόγο. Σήμερα το Κοινοβούλιο έχει βραβεύσει πλέον ε, με το βραβείο Ζαχάροφ 2019 τον κύριο Τότι. Ο κύριο Τότι είναι επικεφαλή, είναι μάλλον ένα έγκριτο οικούρο, ε, οικονομολόγο και διανόμενο, και έχει απλώ αγωνιστεί για την ειρήνη και τα δικαιώματα των Ουγγούρων. Έχει καταδικαστεί σε ισόβια και δεν μπόρεσε να έρθει στο Στρασβούργο να αναλάβει το βραβείο του βεβαίω. Σήμερα και αυτές τις μέρες εκπροσωπήθηκε εδώ από την γενναία κόρη του, την Γέβεν. Και εδώ ζητούμε την άμεση και την απευθείας απελευθέρωσή του. Ε, η περιοχή της Ξενγιάνγκ έχει γίνει μια αιστεία μαζικής ε, παρακολούθησης εθνοτική ε, θρησκευτική φιλετικής, κοινωνική δίσδυση. Κάθε πτυχή του κοινωνικού βίου παρακολουθείται. Οι Ουιγούροι επιχρόνονται να παρνηθούν τη θρησκευτική σκεφτική και πολιτιστική του ταυτότητα στα λεγόμενα στατόπεδα ε, αναμόρφωση. Η Κίνα έχει δεσμευτεί όμω να ακολουθεί στο πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων όπω και παγκοσμίω. Έχουμε καλέσει την κινέζικη κυβέρνηση να απελευθερώσει όλου του κατουμένου εφόσον ε, δεν υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Θα πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα στρατόπεδα και οι ε, δράστες παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προσέλθουν ε, ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει στοχευμένες κυρώσεις κατά των υπετίων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ο κύριος Μπένιον για δύο λεπτά για τους Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάνω από δύο δεκαετίε ο Ιλάν τότε έχει εργαστεί άοκνα για να υπάρξει διάλογο και κατανόηση μεταξύ Ουιγούρων και τη κεντρική κοιναζική κυβέρνηση. Όμω καταδικάστηκε το Σεπτέμβριο του 2014 σε ισόβια για τι προσπαθίε αυτέ. Ε, και μετά από μία ψευδοδίκη δύο ημερών. Ε, σήμερα έλαβε πλέον το βραβείο Ζαχάροφ φέτο και είναι ο νέο βραβευτή. Όμω δεν είναι ο μόνο που αποφέρει λόγω του κινέζικου καθεστώτο. Υπάρχουν και άλλοι, ε, Ουιγούροι, οι έχουν ε, υποβληθεί σε ανίποτα βασανιστήρια από, από την κοινωνική κυβέρνηση την τελευταία διετία. Λόγω τη μοναδική θρησκευτική και εθνοτική του ταυτότητα. Από τον Απρίλιο του 2017, πάνω από ένα εκατομμύριο αθώοι Ουιγούροι έχουν αυθαιρέτω συλληφθεί και καταδικαστεί σε τόπεδα αναμόρφωση. Πρέπει να απαρνηθούν την εθνοτική του ταυτότητα, τη θρησκεία του και να δηλώσουν την πίστη του στην κοινωνική κυβέρνηση. Πραγματικά ανησυχώ ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει η κινέζικε αρχέ να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι ελευθερίε. Θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσει για τι παραβιάσεις αυτών. Η κινέζικη κυβέρνηση πρέπει αμέσω να πάψει τι αυθαίρετε αυτές συλλήψει και φυλακίσει, να κλείσει όλα τα στατόπεδα, ε, τα κέντρα ε, φυλάκισης και να απελευθερώσει του κρατουμένου. Ταυτόχρονα θέλουμε οι κινέζικες αρχές να επιτρέψουν ελεύθερη πρόσβαση ε, στην περιοχή τη Ξινγιάνγκ, την αυτόνομη περιοχή αυτή, για του δημοσιογράφου και του διεθνεί παρατηρητέ. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς και να συνεχίζουμε να έχουμε κανονικές σχέσεις με την Κίνα ενώ υπάρχουν αυτές οι ε, φρικτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά την άποψή μου, έχουμε τις σοβαρότατες παραβιάσεις στην περίπτωση αυτή ε, παγκοσμίω σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ελπίζουμε ότι η απόδοση του βραβείου στον κύριο Τότη θα οδηγήσει στην απελευθέρωσή του και ότι εφ' εξής θα επιτρέψει να υπάρξει και αλλαγή στην ε, στρατηγική, την στάση των κινέζικων αρχών στην, ε, απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Μπίτικοφερ για δυόμιση λεπτά για τους πρασίνους. Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Μπορέα για τα σταράτα λόγια σας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική του κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος κατά των δεν ποτέ ήταν φιλελεύθερη. Αλλά το 2014 ε, έγινε μια αυταρχική στροφή στο Ξιν που δημιούργησε το χειρότερο αστυνομικό κράτος παγκοσμίως σήμερα. Αυτή η ακραία πολιτική γνωρίζει και μια εσωτερική αντίθεση, όπως μάθαμε από τα τηλεγραφήματα για την Κίνα, China Cables. Μια τόσο μεγάλη χώρα με τέτοιο μακρύ ε, πολιτισμό, μακροχρόνιο, είναι ντροπή να εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μεν απαραίτητη, αλλά δεν είναι δικαιολογία για να καταπολεμούν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν σκέφτονται όπως οι Κινέζοι που, δεν λατρεύουν το Θεό τους όπως θέλουν οι Κινέζοι και που δεν μιλούν όπως θέλουν οι Κινέζοι. Έχει έρθει η ώρα να σταματήσουν τα ψεύδη και οι δικαιολογίε και ε, οι παρελκυστικές κινήσεις και να κλείσουν αυτά τα στρατόπεδα. Εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πέρα από τα επικριτικά μας σχόλια. Γι' αυτό το κοινοβούλιο μας ζητεί να σταματήσουν οι εξαγωγές και η μεταφορά τεχνολογίας, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για να ενταθεί η κυβερνό παρακολούθηση. και δεν θα πρέπει τα προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία σε τέτοια στρατόπεδα συγκέντρωσης να εξάγονται προς την Ευρώπη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να απαγορευθούν από τις ευρωπαϊκές αγορές. Καλούμε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες να χαράξουν σαφείς κόκκινες γραμμές. Κινδυνεύει η φήμη τους αν δεν το κάνουν και αν δεν εφαρμόσουν ε, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην ενέχονται σε τέτοιες κατασταλτικές πρακτικές. Και αυτό που χρειαζόμαστε επίσης είναι ένας μηχανισμός κυρώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το έχετε συζητήσει με τους Υπουργού Εξωτερικών, κύριε Μπορέλ, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και μάλιστα γρήγορα να γίνει. Και μια τελευταία πρόταση για τον Ήλαμ Τότι. Ε, το βραβευθέντε σήμερα με το βραβείο Ζαχάροφ. Δεν τον αφήνουν να δει την οικογένειά του. Δεν την έχει δει την τελευταία διετία. Ακόμα και αν αυτό το εγγυάται η κινέζικη νομοθεσία. Θα πρέπει όλοι να επιμείνουμε. Η οικογένειά του θα πρέπει να, να, να, επιτρέπεται να γνωρίζει πού διαβεί και πού, πού είναι ο άνθρωπος αυτός και να τον δει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπονφρίσκο από την ομάδα ID για δύο λεπτά. Κυρία Πορφίσκο, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, είπατε πρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μακρός ο δρόμος του μεταξύ. Ο 73% του παγκόσμιου πληθυσμού στο μέλλον. Η Κίνα αυτή τη στιγμή εφαρμόζει δικούς της κανόνες για τους πολίτες. Και για την περιοχή των Ουιγούρων ένα από τα βασικά κομβικά σημεία του φιλόδοξου εγχειρήματος της Κίνας 100 ε, δολαρίων βρίσκεται, γίνεται το τέλειο άλοθη για να καταστήλουμε σήμερα την ε, επιθυμία αυτοδιάθεσης του τοπικού πληθυσμού. Ο νέος δρόμος του μεταξιού λοιπόν μπορούν, ε, μπορεί να γίνει ένας δρόμος για τα εμπορεύματα αλλά απαγορεύει τα δικαιω... τη δημοκρατία και τα δικαιώματα φαίνεται. Ε, θεωρώ επίσης ε, είπατε εκπρόσωπε, ότι η πολιτική γειτονία θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει γεωπολιτικών παραμέτρων που να ισχύουν ε, διεθνώ, όχι μόνο γεωγραφικών όρων. Η παγκόσμια η ιστορία και η παράδοση των Ουγγούρων δείχνει ότι ε, η χώρα η περιοχή αυτή είναι θύμα του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου. Ε, έχει γίνει τίμημα στο βωμό της επέκτασης και της ξέφρενης ε, υπεροχής ε, της τεχνητής ευθείας και του εμπορίου της. Οι μηχανισμοί της κοινωνικής πίστοσης, η πώληση συγκινήσεων και συναισθηματών επιτρέπουν τη μαζική παρακολούθηση 1,5 δις ανθρώπων ε, με την ε, κυβέρνηση του Πεκίνου να παρακολουθεί με τα big data ό,τι θέλει, αλλά με καλές εμπορικές συναλλαγές, με τεράστιες βάσεις δεδομένων, όπου σειραίουν τα προσωπικά δεδομένα όλων των πολιτών, βάσει ενός κεντρικά οργανωμένου συστήματος που δεν κάνει διάκριση μεταξύ ιδιωτικού βίου και δημόσιου. Ε, εδώ λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση απαράδεκτη. Η Ευρώπη με τις θεμελιώδες τη αξίε δεν μπορεί πλέον να δεν μπορεί απλώ να λαμβάνει γνώση. Πρέπει να σκεφτούμε ότι γρήγορα ο Ιγούρι θα γίνουμε όλοι μα. Ευχαριστούμε. Επόμενη κυρία Φωτίγκα για 1,5 λεπτό για του συντηρητικού και αναρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Παρά τα πειράματα στον τομέα της οικονομίας, η Κίνα παραμένει ένα κομμουνιστικό κράτος που μαζικά εκφοβίζει μεγάλες ομάδες της ίδιας της, της κοινωνίας. Από το Νοέμβριο του 2019 διέρευσαν τα λεγόμενα China Cables. Από τότε λοιπόν που έγινε αυτό, ο εκφοβισμός στην αυτόνομη περιοχή Ξινγκιανγκ, ε, εκεί που ζουν οι Ουιγούροι, έχει γίνει πιο ξεκάθαρη σε εμάς. Φυσικά, τα στρατόπεδα κράτησης δεν είναι χώροι εθελούσιας εργασίας. Φυσικά, υπάρχει μαζική παρακολούθηση με όλα τα τεχνικά μέσα. Επιζητούμε αποφασιστική δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, πραγματικά πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι από την πλευρά μας. Κάνω έκκληση λοιπόν να κλείσουν αυτά τα στρατόπεδα, να υπάρχουν στοχευμένες κυρώσεις έναντι εκείνων που είναι υπεύθυνοι ε, ε, δράστες, δηλαδή αυτού του εκφοβισμού. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ε, Γκουε για ένα λεπτό η συνάδελφος Βιρανέλα Βαρούιχ. Ανησυχούμε από όσα μαθαίνουμε από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ξινγιάν και από τα κινέζικα τηλεγραφήματα, China Cables. Θα πρέπει να βρούμε ε, ποιος έχει την ευθύνη. Η ομάδα μας ανέκαθεν είναι κατά της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων απανταχού της γης. Και θα πρέπει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία να προστατεύεται, γιατί βλέπουμε ε, εκτροπές και ολισθαίνουμε προς ε, αυταρχικά καθεστώτα. Θα πρέπει ε, σε πολυμερή φόρα να συζητούμε. Γι' αυτό μιλάμε για κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τις οποίες καταγγέλουμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι ο καταλληλότερος τέρος για να μιλήσει για περιστολή των ελευθεριών. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τόσο εμπορικό πόλεμο, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι και άλλε κυρώσει, αλλά διάλογο, πολυμερή συνεργασία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ στο Κοινοβούλιο συχνά χρησιμοποιούμε τα θεμέλια δικαιώματα ως εργαλείο για γεωπολιτικές επιθέσεις. Και σήμερα που είναι η μέρα του μετανάστη, θα ήθελα ως Ευρωπαία να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Και να θυμίσω κάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι παράνομος ή λαφραίος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν μπλε κάρτες όταν μιλούν οι εκπρόσωποι εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Καστάλντο. Μη εγγεγραμμένος για ένα, μισή λεπτό. Grazie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φανταστείτε μια κοινωνία όπου η τεχνητή ευθεία χρησιμοποιεί αυτόματους αλγορίθμους και την αναγνώριση προσώπου για να αποφασίζει ποιο πρέπει να συλληφθεί και να πάει σε ένα στατόπεδο αναμόρφωσης. Οι φοιτητέ, που στην πραγματικότητα είναι κρατούμενοι, δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Βρίσκονται διαρκώς από παρικολούθηση και πρέπει να μαθαίνουν ε, κινέζικα, μανταρινικά και βεβαίως ε, πρέπει να παρνηθούν την ταυτότητά τους και να γίνουν Κινέζοι. Πρέπει ε, να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν το υπόλοιπο της ζωής τους και το καθεστώς το οποίο θα ζουν. Μιλάμε για μια ε, τραγωδία. Κάτι έχει πάει στραβά. Η ανθρωπότητα κάποια στροφή πήρε λάθο. Ε, ε, σήμερα το 2019 στην Ξινγιάν ε, πάνω από ένα εκατομμύριο Ουιγούροι βρίσκονται σε αθαίρετη κατάσταση σύλληψη και πρέπει να απενεθούν την ταυτότητά του γιατί του έχει κρίνει επικίνδυνο στο κομμουνιστικό καθεστώ τη Κίνα. Θέλουμε αυτομάτω κυρώσει για τι ε, απαράδεκτε, τι ασύλληπτε αυτέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πάψουν οι εξαγωγέ τεχνολογικών μέσων που επιτρέπουν αυτό το profiling και πρέπει αυτή τη δυσάρεστη πραγματικότητα των κινέζικων αρχών να την αναγνωρίσουμε. Πρέπει να ε, αναλάβουν τι ευθύνε του οι Κινέζοι. Η δική μας, ε, το δικό μα ανάστημα των ανθρωπίνων όντων θα κρυθεί από την δυνατότητά μα να μετρηθούμε με αυτήν την κρατική βία. Όπω έκανε ο Ιλάμ ε, τότε και ε, ο οποίος πλήρωσε τις συνέπειες της αντίστασής του, αλλά εγώ ε, στήριξα την υποψηφιότητά του ε, από πλήρη αποφασιστικότητα, διότι είμαι πεπισμένος ότι είναι ηθικό μας καθήκον να αγωνιστούμε συμπαρατασσόμενοι με αυτούς τους ακτιβιστές, προασφιστές της ελευθερίας. Ελπίζω σύντομα να απελευθερωθεί και να ξαναβρει την κόρη του. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, παρακαλούμε, σκεφτείτε λίγο και τους διερμηνείς όταν επιταχύνεται. Επόμενος ο κύριος Γκάλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο και Πατεκπρόσωπο κύριο Μπορέ για τα όσα είπε στην ερεκτήρια ομιλία του και Βεβαίω, ε, αν ήταν παρόν και στην απονομή του βραβείου Ζαχάροφ, θα παίρναγε και ένα διαφορετικό πολιτικό μήνυμα. Ένα πολιτικό μήνυμα που πρέπει να ε, ξεκινήσει από το σώμα αυτό. Διότι όλοι θα πρέπει να επικρίνουμε την κατάσταση στην Ξυγιά και είμαστε όλοι εδώ ομόφωνα σύμφωνοι. Ε, έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Πιστεύω ότι όσα λαμβάνουμε ω ειδήσει από τι πρεσβείε μα είναι σαφή ε, πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα όπως προβλέπονται στο Σύνταγμα ε, και πρέπει διεθνώς να σεβαστεί η Κίνα όσα έχει υπογράψει, τα οποία θα πρέπει και να κυρωθούν. Και μετά θα πρέπει οι υπεύθυνοι του ΟΗΕ, οι πετετραμένοι, να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την περιοχή για να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Ε, ε, η Κίνα είναι ένα μεγάλο κράτος το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζει έτσι μια μικρή μειονότητα. Οι Ουιγούροι δεν απαιτούν τίποτα διαφορετικό ε, από το δικαίωμα να είναι αυτόνομοι ως πληθυσμός. Και γι' αυτό έχουν την πλήρη υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κεπχάρτ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα κινέζικα τηλεγραφήματα και μας έδειξαν ε, ε, πώς ε, δρά η κυβέρνηση και πώς θέλει να εξορροθρεύσει την ταυτότητα των Ουιγούρων και μάλιστα ανερυθρίαστα. Είναι οι χειρότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζούμε. Περιμένω από σας κύριε Μπορέλ και τα κράτη-μέλη να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που έχετε ήδη κάνει. Ε, ε, να τα λέτε έξω από τα δόντια ε, στους Κινέζους και στην κυβέρνησή τους. Αγωνιστείτε για να κλείσουν αμέσως αυτά τα στρατόπεδα αναμορφωτήρια και να ανοίξει η περιοχή ε, ε, για να ε, μεταβούν εκεί ανεξάρτητοι παρατηρητές να μας πούν τι γίνεται. Υπάρχουν και διεθνείς εταιρείες στην Ξινγιάνγκ και ζητούμε να εξετάσετε κατά πόσο συμμετέχουν σε αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιστοίχω να υπάρξουν και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε τέτοια προϊόντα που να παράγονται από καταναγκαστική εργασία και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην βρίσκουν το δρόμο του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχουν πρόσβαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία είναι να τονίζουμε συνεχώ και ομόφωνα ότι η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου ε, είναι αναπαλωτρίωτες ε, προϋποθέσεις για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νετβέλτ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Παπτέκ. πρόσωπε. Σας θυμάμαι στην άλλη θέση εδώ πάνω στο πόντιου πριν από μερικά χρόνια αυτή εδώ η υπόθεση θα είναι η βασική διαλήθος για την νέα γεωπολιτική επιτροπή. Πριν από μερικά μερικές ε, μέρες ε, υπήρξε από μια γυναίκα η διαρροή αυτών των China Cables μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα τέτοια εργαλεία η Κίνα επιδεικνύει την απολυταρχική της στάση. Αυτά τα εργαλεία αν υπάρχουν ε, μπορούν και χρησιμοποιούνται. Σήμερα δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ στον Ήλαμ Τότι ως πολιτικό μήνυμα για το που βρίσκεται η Ευρώπη. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που δίνουμε το βραβείο Ζαχάροφ σε μαχητές της ελευθερίας στην Κίνα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η απέτηση να απελευθερωθούν οι Ουιγούροι που κρατούνται στα στρατόπεδα, γιατί αυτό είναι. Άκουσα πολλές καλές συστάσεις από τους συναδέλφους για το πώς θα προχωρήσουμε, όμως υπάρχει και ένα νέο εργαλείο ε, στην πρότασή μας που είναι το ευρωπαϊκό, ο Ευρωπαϊκός Νόμος ε, που πρότεινε ε, το Συμβούλιο. Θα γίνει πραγματικότητα αυτό χωρίς καθυστέρηση. Θα προσπαθήσετε να ψηφιστεί ε, με τρόπο που να μην μπορεί καμία χώρα να ασκήσει βέτο. Θα διασφαλίσετε ότι η ΜΚΟ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ε, Κοινοβούλιο και τα άλλα κοινοβούλια θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Θα μπορέσει η Ευρώπη να γίνει μια νέα γεωπολιτική υπερδύναμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Γκρεγκόροβα για ένα λεπτό έχει το λόγο σε επόμενη ομιλήτηρια. Κύριε Μπορέλ, μιλάμε για τις πρόσφατες διαρροές ε, που αποκάλυψαν ότι οι Κινέζοι ε, πρέσβησε και υψηλά στελέχη της κυβέρνησης ε, κρύβουν από εμά τη μαζική πολιτιστική γενοκτονία που διαπράττεται αυτή τη στιγμή Κίνα, στην Κίνα. Χθες ε, συναντήσαμε την κόρη του κυρίου Ιλαμπτότη. όμως τον ίδιο δεν μπορέσαμε να το συναντήσουμε γιατί είναι κλειδωμένος μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης εκεί μέσα εδώ και δύο χρόνια ε, των ε, τυραννούν θέλει ε, η κόρη του να είναι στην Κίνα, να είναι μαζί και ασφαλής. Την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η γενοκτονία, στη χώρα μου ο πιο ε, ισχυρός και πλούσιος άντρας ε, χειρίζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για επιχειρηματικούς λόγους. Ε, ζητώ συγγνώμη, αν ήμασταν και εμείς ε, στην Κίνα και κάναμε μια τέτοια ομιλία θα μπαίναμε κι εγώ και η οικογένειά μου π.χ. Ε, σε ένα τέτοιο στρατόπεδο. Εμείς συνάδελφοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων κατά της δικτατορίας της Κίνας, ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οικονομικές κυρώσεις. Κύριε Μπορέλ, πρέπει να δράσετε αμέσως. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κοράου για ένα λεπτό είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά είναι απαράδεκτα παρά τις συνεχείς εκκλήσεις από την διεθνή κοινότητα και τις πρόσφατες δημοσιεύσεις εγγράφων που στην ουσία αποδεικνύουν τις επονίδιστες αυτές πράξεις στην ε, αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων, η κινέζικη κυβέρνηση φαίνεται ότι ε, παραμένει αδιάφορη και συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε μια χώρα σαν την Κίνα η οποία συνεχώς θέλει να την βλέπουμε ως έναν αξιόπιστο συνομιλητή στο παγκόσμιο πεδίο ε, αυτή η σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι αποδεκτή. Επίσης, συνεχίζει την δίωξη των Ουιγούρων και άλλων μειονοτήτων εκτός των εθνικών της συνόρων. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και να λάβουμε αντίμετρα. Είπαμε πράγματα στον καθηγητή Λαμπτότη. Ε, αυτά που του είπαμε δεν αφορούν μόνο αυτόν, αλλά όλους τους Ιγούρους πολίτες ε, που μάχονται στην ίδια μάχη. Ως Ευρωπαίοι λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα της μειονότητας των Ιγουρών στην περιοχή Σινγκιάνκα και σε όλες τις χώρες των Εθνών. Αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να δοθεί μόνο στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχουμε κοινέ προσπάθειες για να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Έχω μια σύγχυση τώρα. Ως προς ε, το αν είχατε εξαντλήσει το χρόνο σας, ελπίζω να μην σας διάκοψα ως μειόφυλλα. Ο κύριος Μακάλιστερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αυτά που μαθαίνουμε για τους Ιγούρους και άλλες μειονότητες ε, στο Xinjiang μας ανησυχούν πολύ. Τι έχει σημασία τώρα. Τα, ε, να, οι αυθαίρετες συλλήψεις χωρίς απαγγελία κατηγορίας θα πρέπει να τερματιστούν αμέσως και οι κρατούμενοι να φεθούν ελεύθεροι άνευ όρων. Δεύτερον, οι αρχές του Πεκίνου θα πρέπει ε, να αφήσουν να πάνε στο Τζινγκιάνγκ ε, δημοσιογράφοι ε, και παρατηρητές ανεξάρτητοι και η Επίτροπος τη αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ και οι κρατούμενοι από το Ξινιάνκ να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Είχαμε την 21η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα. Διατράνωσαν και οι δύο ότι όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα είναι ε, ενιαία, πανανθρώπινα και οικουμενικά. Καλείται η Κίνα όλα αυτά να τα εφαρμόσει. Καλωσορίζω τα σαφή σας λόγια κύριε Μπορέλ, αλλά και το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε αύριο το μεσημέρι. Ιδιαίτερα ε, η ε, έκκληση για στοχευμένες κυρώσεις είναι αυτή που με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ κυρία Σάντος. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε η Κίνα συνεχίζει την πολιτική συστηματικής παραβίασης και έλλειψης σεβασμού για τα βασικότερα δικαιώματα του πολίτη. Η στάση αυτή αποδεικνύεται με τις εναρρύθμιστες υποθέσεις πολιτών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο ή με την απαράδεκτη κατάσταση στην Ξινγιάν και το Θιβέτ. Πραγματική πολιτιστική γενοκτονία. Ε, ένα στοιχείο που αποδεικνύει αυτή την πολιτιστική ισοπαίδωση είναι ότι η κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ιγούρων, ακριβώς η ίδια κυβέρνηση που ε, ήθελε να γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια ερήνευση στο Θιβέτ. Τελείως υποκριτική, διπρόσωπη για όσα συμβαίνουν και συνεχίζονται. Η αναμόρφωση, η πολιτιστική αναμόρφωση, τα βασανιστήρια, τα αστυνομικά έργα. Η ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτά. Πρέπει επιτακτικά να πετήσουμε την άμεση και άνεφόρον απελευθέρωση του Ιλάμ τότε και όλων των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, ε, και να πάψει η εισαγωγή από προϊόντα που είναι προϊόν των καταναγκαστικών έργων. Πρέπει να υπάρξουν στοχευμένε κυρώσει ώστε να πιεστεί η κινέζικη κυβέρνηση να κλείσει αυτά τα στρατόπεδα και να δώσει τέλο στι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κιουτσούκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Μπορέη. Η συζήτηση αυτή δεν έχει σκοπό να στραφεί κατά τη Κίνα ή τη κινέζικη κυβέρνηση, αλλά να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα προστατεύσουμε. Θέλω να αποτύσω ειδικό φοροτιμή στον Ιλιάμ Τότι, ο οποίο έλαβε το βραβείο Ζαχάροφ σήμερα. Είναι ένα γνωστό ε, ε, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διανοούμενο και υπερασπιστή τη κοινότητα των Ουιγούρων. Επί 20 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκε διαλόγου για να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μεταξύ Ουιγούρων και των, Χαν, των Κινέζων ε, Χαν. Ε, ε, καταδικάστηκε όμως σε φυλάκιση το 2014 και έκτοτε βρίσκεται πίσω από τα σίδερα. Κύριε Μπορέι, πραγματικά ε, ζητώ αμέσως να απελευθερωθεί από τη φυλακή ο κύριος Μπορέι, ο κύριος ε, Τότη, συγγνώμη, και να σταματήσουν ε, οι παραβιάσεις κατά των Ουιγούρων στην Κίνα. Ευχαριστούμε. Φων Κραμόν Ταουμπαντέλ από τους Πρασίνους. Thank Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, είπατε εκπρόσωποι. Ε, Είδαμε, ο, αν ακούσουμε τις ειδήσει από την Κίνα, θα πιστέψουμε ότι όλα πάνε καλά. Ε, Όμω οι Κινέζοι είναι αδύναμοι, διότι ξέρουν ότι αυτά που κάνουν με τους, εναντίον των πολιτών του είναι στην πραγματικότητα ε, εντελώ ε, ανήθικα. Είναι απαράδεκτα οι καταπιέσει, η παρακολούθηση και η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κινέζικη κυβέρνηση γνωρίζει ότι παραβιάζει όλου του κανόνε και τι διεθνεί συμφωνίε. Έχει αναλάβει ευθύνε να προστατεύσει του πολίτε τη η Κίνα και δεν το κάνει. Είναι δική τη ευθύνη να κοιτάζει το καλό των πολιτών τη. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι τα ελάχιστα πρότυπα ισχύουν και στην Κίνα. Εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να σώσουμε του Ουιγούρου στην Κίνα εάν δεν είμαστε ενωμένοι εάν δεν ενώσουμε τι δυνάμει μα. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και να καλέσουμε την Κίνα να αναλάβει ευθύνε. Χωρί μια ε, κοινά συμπεφωνημένη στρατηγική δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη ζωή όσων είναι στην Κίνα. Όμω δεν είναι μόνο οι κυβερνήσει και οι πολιτικοί ηθήνοντε που πρέπει να ακολουθήσουν τον κοινό αυτό δρόμο και τα όσα θα συμφωνηθούν βάσει μια στρατηγική για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και εταιρείε, επιχειρήσει που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται αλλά δεν ξέρουν τι βγάζουν στην Κίνα και στην Ξινγκιάν. Οπότε, χωρί Εκείνε δεν θα πετύχει η στρατηγική μα. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Ζόφκο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, η πρόσφατη ιστορία μα δείχνει ότι οι ε, θρησκευτικές μενότητες συχνά υποφέρουν ε, και παραβίζονται τα δικαιώματά τους. Όταν αυτό συμβαίνει κάπου στον κόσμο, αυτό ω ε, ντόμινο έρχεται και φέρνει επιπτώσει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Τα όσα συμβαίνουν με του Ιγούρου στην Κίνα είναι επίκαιρα και καλωσορίζω τη συζήτηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Κοινο... Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να κοιτάξουν τι συμβαίνει με την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών και την απονομή του βραβείου Σάχαροφ στον κύριο Τότη, ο οποίο ε, συστηματικά προασπίζεται τα δικαιώματα των Ουιγούρων. Πρέπει να κοιτάξουμε αυτήν την τάση που έχει αυξητική πορεία για να παρα... καταπιέζονται οι μειονότητε και να διώκονται παρομοίω και αλλού, όπω οι χριστιανοί στην Πουρκίνα Φάσο. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στην τελευταία σύνοδο στο Στρασβούργο συζητήσαμε τη δίωξη καθολικών και προτεστάντων στην Αλγερία. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανεξιθρησκεία ε, και η ελευθερία είναι η ακρογωνία λύθη μια ελεύθερη και δίκαιη κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή του διαθρησκευτικού διαλόγου ε, στι ανακοινώσει τη στρατηγική του και προκειμένου να υπάρξει μια διάσταση συμφιλίωση και στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Κλουξμάν για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν διαβάζεις το Κοράνι, σε περιμένει στρατόπεδο. Αν έχεις μουσεί, σε περιμένει στρατόπεδο. Στέλνεις ευχές σου για τη μουσουλμανική γιορτή, για τον Μπαϊράμι, πας στο στρατόπεδο. Αυτά παθαίνουν οι Ουγγούροι αυτή τη στιγμή και οι μεγάλες σιωπές επιτρέπουν τα μεγάλα εγκλήματα. Οφείλουμε να πούμε ότι ο κόσμος ε, αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχει σιωπήσει. Εμείς πάσαμε αυτή τη σιωπή δίνοντας το βραβείο Ζαχάροφ στον Ιλάμ τότε. Δεν φτάνει αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα και κυρώσεις κατά των Κινέζων ηθινόντων που ενέχονται άμεσα σε αυτό που σήμερα συνιστά τη μεγαλύτερη πολιτική μαζικού εγκλισμού παγκοσμίω. Χρειάζονται κυρώσεις και κατά των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Και τέλος, οι ευρωπαϊκές εταιρείες να εφαρμόσουν ε, το καθήκον επαγρύπνησης, ιδιαίτερα οι κλωστοεφαντουργικές ας πούμε να μην επωφελούνται από αυτό που σήμερα είναι μια παράδεκτη πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπερνάχ Γκετά. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Μπορεί κανείς να τους αποκαλέσει όπως θέλει και τα ε, αναμορφωτήρια, στρατόπεδα αναμόρφωση που λέει το Πεκίνο, αλλά ένα στου εννέα Ουιγούρους, ένα εκατομμύριο είναι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ε, ε, θα πρέπει εμείς να γανακτούμε, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να θυμίσουμε στους Κινέζους ηθήνοντες ότι δεν νοείται πραγματική ισχύ χωρί ευθύνη. Ο κόσμος χρειάζεται την Κίνα, γιατί χωρίς εκείνη δεν υπάρχει η ελπίδα να φύγει η αναρχία από τη διεθνή σκηνή και να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις χωρίς τις δεν υπάρχει σταθερότητα. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε στους Κινέζους συνθήναντες. Αλλά ε, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει ούτε εσωτερική ειρήνη ούτε διεθνής ασφάλεια. Ας ε, λοιπόν όσο σοφή έχει αποδειχτεί η ιστορία σας των χιλιάδων ετών. Κλείστε τα στρατόπεδα, αφήστε τους λαούς σας να αναπνεύσουν και αφήστε ελεύθερο και τον Ιλάμ Τότι. Ευχαριστώ πολύ. Νταβίτ Λέγκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που στοχεύονται και διώκονται λόγω των πεπιθήσεών τους. Ξέρουμε ότι τους γονείς τους χωρίζουν από τα παιδιά. Καταστρέφονται οι οικογένειες. Ξέρουμε επίσης ότι τα πολιταρχικά καθεστώτα κρατούν εκατομμύρια ανθρώπους στα λεγόμενα στρατόπεδα αναμόρφωσης, τα οποία μας φέρνουν ε, φρικτές μνήμες για παρόμοια στρατόπεδα που είχαμε στην πρόσφατη ιστορία μας στην Ευρώπη. Ήμασταν πολύ αργοί στην αντίδρασή μας έναντι του, των φρικτών κλιμάτων της κινέζικης κυβέρνησης. Φίλοι, συνάδελφοι, είναι η στιγμή να σταματήσουμε να μασάμε τα λόγια μας ε, για την Κίνα και το κομμουνιστικό της καθεστώς. Ε, το βραβείο Ζαχάροφ στον Ήλαμ τότε δείχνει ότι δεν θα δεχτούμε πλέον τα εγκλήματα της Κίνας κατά των Ουιγούρων. Αύριο έχουμε την, ε, το ψήφισμα για τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις για τις μαζικές κρατήσεις των Ουιγούρων. Ας υποστηρίξουμε τους Ουιγούρους όμως όχι μόνο με κυρώσεις γιατί θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες κάθε φορά που απειλούνται και αυτό είναι που ε, σηματοδοτεί την Ευρώπη και δεν πρέπει να το αφήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο λόγος Πηγαίνει στην κυρία Τζιλ ένα λεπτό. Κύριε, είπατε εκπρόσωπο, καλώς ήρθατε ξανά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στην αίθουσα, σε αυτό το σώμα, με το νέο σας ρόλο. Αντιμετωπίζουμε μία από τις μεγαλύτερες